δηλαδή τα αποθέματα Ρέγκας στα δυτικά της Σκοτίας. Και μια και πρόκειται για Σκοτία, αρμόδιος συγητής είναι ο κύριος Στρούαν Στίβενσον. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Δανική Προεδρία πριν από μερικές εβδομάδες με ενημέρωσε ότι δεν θα έχουμε ε, συμφωνία πρώτη ανάγνωση επί της έκθεσης μου για το πολιτέ ε, σχέδιο για το απόθεμα Ράγκα στα δυτικά της Σκοτίας. Έχουμε παρόμοιο ε, μπλοκάρισμα και τη έκθεση Πάντε Κόμπ Γκάλαχερ του πολιετούς σχεδίου για το Σαβρίδι του Βορειοατλαντικού. Τέσσερα χρόνια έχει αποτελματωθεί η κατάσταση και έκθεση Μπιλμπάου Μαραντίκα για το απόθεμα ε, γάβρου στην, ε, στο φυσικό κόλπο επίση έχει μπλοκαριστεί. Δεν είναι θέμα λοιπόν ε, μόνο μια έκθεση. Έχουν μπλοκαριστεί συστηματικά εκθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν υπάρχει αμφισβήτηση για θέματα καταξιδότηση πράξεων ή εφαρμοστικών πράξεων. Το Συμβούλιο φαίνεται ότι αρνείται να αποδεχθεί ότι με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν είναι το μοναδικό αρμόδιο όργανο και δεν έχει το τελικό λόγο για τα θέματα αυτά. Ε, επιμένω ότι στην έκθεσή μου ε, για το πολιτικό σχεδίο απόθεμα Ρέγκα, με βάση τις κατεξουσιοδότηση πράξη θα αξιολογηθούν ε, τα πολιτή προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πλήρη όμω διαβούλευση με το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνηση της Θάλασσας καθώς και της Ειδική Τεχνική, Οικονομική και Επιστημονική Επιτροπή, καθώ και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τα Πελαγικά Αποθέματα. Η εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιηθούν εφαρμοστικέ ε, πράξει, κάτι που θα δώσει περισσότερο λόγο στο Συμβούλιο για την αξιολόγηση του πολίτου σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή όμω, το, το Κοινοβούλιο συγγνώμη, μόνο μπορεί να συμβουλεύσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αγνοήσει αυτή την γνωμοδότηση. Φαίνεται ότι το μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο προ προκλήθηκε από, την ανεπίσημη, από τις ανεπίσημες ομάδες εργασίας και όχι από τους υπουργούς. Φαίνεται ότι οι ομάδες εργασίας κατέσαν ομήρου με βάση το άρθρο 43.3 της Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα πολίτη σχέδια, γιατί ε, αποκτούν έτσι τη μοναδική αρμοδιότητα. Το Συμβούλιο και. Συγγνώμη, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεκδικούν το άρθρο, την εφαρμογή του άρθρου 43.2 ε, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου συμφωνούν με την ερμηνεία του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Αλλά παρόλα αυτά το Συμβούλιο εμένει πεισματικά στη θέση του για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και συνεχίζεται ε, το μπλοκάρισμα της κατάστασης. Ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινής ε, αλληλευτικής πολιτικής, αυτό το μπλοκάρισμα στην αναμοθετική διαδικασία είναι πολύ επικίνδυνο. Δημιουργία στάθεια στην αγορά, και δεν δίνει στους αλληλείς και στους μεταπιτές την απαραίτητη ασφάλεια που απαιτείται για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Τα πολιετή σχέδια διαχείρισης θα πρέπει να εφαρμοστούν για τα βασικά εμπορικά είδη. Πώς μπορούμε να επιχειρηματολογούμε ότι δεν υπάρχουν κονδύλια στο Ταμείο Αλίας και Θάλασσας για να χρησιμοποιηθούν για την εξυγχρονισμό των αλληλευτικών σκαφών όταν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε στους ελίες μας ε, την ε, διαβεβαίωση ότι μπορούν να δανειωθούν από τις τράπεζες για να εξυγχρονίσουν τα αλληλευτικά του σκάφη με βάση την βεβαιότητα που θα έχουν από τα πολιτή σχέδια διαχείρισης αποθεμάτων. Γιατί με την κρίση ε, ε θα μπορέσει ο ο Αλίας να αναλάβει τον κίνδυνο και να στη 2 εκατομμύρια για να ξεχρονίσει το ελευτικό του σκάφο αν δεν έχει τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχουν πολίτη σχέδια για να εγγυηθούν την δυνατότητα αλίας για πολλά χρόνια. Χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση τη αλίας, να μην προσφύγουμε στα δικαστήρια για να επιληθεί αυτή η κρίση του μπλοκαρίσματος, γιατί αυτή η προσφυγή φαίνεται όλο και πιο πιθανή, αλλά έτσι θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο η μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Ας μην ξεχνούμε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για μια νέα μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής μετά την 1η Πρώτου 2014. Οπότε είναι θεμελιώδου σημασία να επιλύσουμε αυτό το θέμα του μπλοκαρίσματος στο Συμβούλιο και προσβλέπω στην Κυπριακή Προεδρία να ταρακονίσει το Συμβούλιο προκειμένου να σταματήσει αυτό το νομοθετικό μπλοκάρισμα και αυτό το νομοθετικό αδιέξοδο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Επιτροπός Δάλη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Στίβενσον και την Επιτροπή για την εργασία του στην πρόταση αυτή η οποία ευθυγραμμίζει την αλληλεία της Ρέγκας στις ακτές της Χωτίας με την συνθήκη της Λισαβόνας σε συνένεση και συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και ε, του Συμβουλίου αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ότι το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξασκήσει τον ρόλο του και η Επίτροπος κυρία Δαμανάκη είπε ότι τα προγράμματα θα πρέπει να υιοθετηθούν με τακτική νομοθετική διαδικασία. Θέλω επίσης να προσθεθούν παράμετροι ε, ε, στο πρόγραμμα της επιστήμης για όλους κατά τρόπον ώστε να μπορεί να αντικατοπτρίζει το πρόγραμμα ανα πάσα στιγμή τις καλύτερες δυνατές προοπτικές. Και εδώ τονίζω ότι σχετικά με τα αποθέματα τα οποία καλύπτονται από το πρόγραμμα οι ε, τροπολογίες του εισηγητή γίνονται αποδεκτής. Όσον αναφορά την ε, εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η τριετής περίοδος γίνεται αποδεκτή αλλά προβλέπεται ένας κύκλος για αναθεώρηση και καλό θα ήταν οι περίοδοι αυτοί να συνάδουν και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτού υιοθετήσει κατεξουσιοδότηση πράξης θα πρέπει να συμβουλευτεί το, την Επιστημονική Επιτροπή και το Αρμόδιο Συμβούλιο. Ε, κατόπιν της συμφωνίας πέρυσι μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, προβεί σε ε, διαβουλεύσεις και να συμβουλευτεί Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων προτού προβεί στη σύνταξη κατεξουσιοδότηση πράξεων εξού και όσον αφορά τη σχετική τροπολογία δεν την δεχόμαστε και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, και την Επιτροπή για την εργασία της και προσλέπω στη συζήτηση που θα έχουμε. Ευχαριστώ. Εκ μέρου των ομάδων τώρα, πρώτα εκ μέρου του ΕΛΚ, για δύο λεπτά, το λόγο έχει ο κύριο Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή κύριο Στίβενσον ο οποίος με την έκθεσή του αντιμετωπίζει και ε, ε, ε, το βασικό θέμα της αλληλευτικής πολιτικής στην Ευρώπη και ε, με το παράδειγμα το οποίο χρησιμοποίησε για τα αποθέματα της ε, Ρέγκας ε, τονίζει το πώς έχει κατάσταση διότι αυτή τη στιγμή συζητάμε την κοινή αλληλευτική πολιτική η οποία πρέπει να καταπτυχθεί για την περίοδο 2014 με 2020 και βλέπουμε ότι όπου υπάρχει ε, ένα απόθεμα το οποίο διατίθεται στον Ατλαντικό με ποσοστώσεις σχετικά με τα λιεύματα και με μεγάλη απόδοση ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, και ε, θέλουμε τα αποθέματα αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον από τις αλλιευτικές μας επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να παραμείνουν εν ζωή και να συμβάλλουν στην οικονομία αλλά τίθεται το ερώτημα οι πόροι που μας διατίθενται στη θάλασσα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά, δεν πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα λιευτικά δικαιώματα, τι θα γίνει με τους αλληλείς οι οποίοι θέλουν να συνταξιοδοτηθούν και έχουν ή δεν έχουν έναν διάδοχο. Ε, μήπως θα πρέπει να υπάρχει συγχρόνως μία περιφερειακή αντιμετώπιση της αλληλείας, να μην επιλύονται όλα τα θέματα από το κέντρο δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο η επιστήμη να επεμβαίνει αλλά θα πρέπει με την πείρα των αλλιέων να μπορέσουμε να συνεργαστούμε πράγμα το οποίο αναφέρεται σαφώς από τον κύριο Στίβενσον και όταν έχουμε τον ορισμό των αποθεμάτων και γνωρίζουμε ποιες είναι οι κινήσεις των αποθεμάτων αυτών τότε θα έχουμε καλύψει το στόχο μας και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κούν. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Γκουίντο Μιλάνα, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στάνφο Στίβενσον για την εξαιρετική εργασία στην έκθεσή του αντιμετωπίζει τα δύο σημαντικά προβλήματα εδώ. Δεν μιλάμε μονάχα για, μια, ε, για ένα απλό σχέδιο διαχείρισης ε, των, ε, της ΕΡΕΝΚΑΣ, αλλά θέλουμε να υπάρχει απόθεμα και για τους μελλοντικού αλληλείς και να υπάρξει μια πολυετής προστασία, καθώς επίσης και μια πολυετής διαχείριση και πολυετής σχεδιασμός. Ε, πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να δεχτεί την ε, θέση που δίνει το, η συνθήκη της ε, Λισαβόνα. Σκέφτεσαι η ώρα που με φωνή πιο σημαντική από αυτήν που διαφαίνεται από την Επιτροπή Αλληλείας να κάνει μια έκθεση για την Ρέγκα που να παίρνει μια πολύ σημαντική θέση για να ξεπερνάει και τις εξακολουθήσεις πράξη Θεωρούμε ότι σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθεί η φυσιολογική διαδικασία. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το θέμα ενέχει και εμπλέκει και άλλους ε, ε, τομείς ε, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη στην μεταρρύθμιση που λαμβάνει η χώρα τώρα αλλά και τη γεωργία και άλλους. Το σημαντικό θέμα είναι ο σεβασμός της επιθυμίας, της βούλησης του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά τώρα, εκ μέρους των Δημοκρατών Φιλελευθέρων, το λόγο έχει ο κύριος Γκάλεχερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Στίβενσον για την προετοιμασία και παρουσίαση της έκθεσης του. Ε, συμφωνώ απολύτως με τις συστάσει ε, της έκθεσης, κυρίως δε την ανάγκη ε, ε να ε, υπάρχει συνήθι τακτική διαβούλευση με του εμπλεκόμενου φορεί. και βεβαίως θέλουμε να υπάρχει μια συστημική διαχείριση του αποθέματος. Ε, θέλουμε να χρησιμοποιηθεί η φυσιολογική διαδικασία, ε, διότι το Συμβούλιο φαίνεται ότι αρνείται κάποιες πτυχές της συνθήκης ε, της Λισαβόνας. Ο Επίτροπος Νταλή λέει ότι πρόκειται για μια συνήθη διαφωνία μεταξύ των θερμικών οργάνων, αλλά εδώ εμείς διαβλέπουμε αφενός μια σημαντική διαφωνία και αφετέρου βλέπουμε ότι τελικά αυτός που χάνει είναι ο τομέας της αλληλείας. Θέλουμε, συμφωνούμε με τη την ε, μακροπρόθεσμη διαχείριση των ε, ε, αποθεμάτων εδώ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κρίση η οποία θα πρέπει να λυθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν φαίνεται ότι θα λυθεί βεβαίως στην παρούσα θητεία, αλλά ελπίζουμε ότι η επικυπριακή προεδρία θα γίνει μια προσπάθεια επί λύσης του προβλήματος είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό το ε, θέμα ε, γιατί η ρέγγα είναι ένα σημαντικό είδος. Ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα... Το σαφρίδι είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ε, είδος και ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη ε, διασύνδεση ανάμεσα στις ε, δύο, στους δύο πληθυσμούς. Θέλουμε να δούμε ότι να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ορισμένοι ηθήνοντες παραμέλησαν, αναγνώρισαν το Κοινοβούλιο στην διαδικασία την νομοθετική μας δημιουργεί ιδιαίτερα ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα. Ε, η θέση του ε, Συμβουλίου ε, δεν οδηγεί σε, καμία, ε, σε κανένα αποτέλεσμα. Ε, δεν ε, βοηθάει στην σωστή και βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων. Βεβαίως εμείς θέλουμε να αφήσουμε τους πληθυσμούς να αυξηθούν. Θέλουμε να υπάρχει αλίευμα και για το μέλλον. Η διαφορά μας δεν είναι με την Κομισιόν, είναι με το Συμβούλιο και ελπίζω ότι χαίρομαι μάλλον που ακούω ότι η Κομισιόν είναι στο Ευχαριστούμε κύριε Γκάλεχερ. Εκ μέρους των Πρασίνων, για 1,5 λεπτό, το λόγο του κύριος Χάττον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η έκθεση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα στην Επιτροπή Αλίας, κάτι που δεν συνηθίζεται για αλληλευτικά θέματα. Συνήθως είναι επίμαχα τα αλληλευτικά ζητήματα. Πάντως, όπως είπε και ο συγητής, ε, θέλουμε με την έκθεση αυτή να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα και τι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γιατί δημιουργήθηκε μια συγκεχημένη και καθόλου ευχάριστη κατάσταση ό,τι αφορά την, τις αποφάσεις για τη διαχείριση αποθεμάτων ε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με αυτή για να ε, μεταρρυθμιστεί η πολιτική και η διαχείριση και να ξεφύγουμε από συγκεντρωτικές μεθόδους που στο παρελθόν μας απογοήτευσαν τα μάλα. Αντί να ε, διαφυλάσσουμε με έμονο τρόπο τις ε, εξουσίες των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να συμβάλλουμε σε αποκεντρωμένη διαχείριση για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους στόχους των αλλαίων. Μόνο η αποκέντρωση είναι χρήσιμη ώστε οι αλληλευτικές χώρες της Ένωσης ε, να μπορούν να συνεργαστούν στις αντίστοιχες υδάτινες λεκάνες για να συντηρούν και να διαφυλάσσουν τα αποθέματα μακροπρόθεσμα. Βέβαια, ε, ισχυρίζονται ότι η συνθήκη της ε, Λισαβόνας εμποδίζει την αποκέντρωση. Η νομική υπηρεσία όμω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει διαφορετική γνώμη. Αποτέλεσμα, η ησύχηση και ε, όλο και περισσότερη συζήτηση και διαξυφισμοί για τα αντίστοιχα δικαιώματα και εξουσίες των θεσμικών οργάνων. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο αυτή την ιδεολειψία και τον προστατευτισμό για τα δικά μας προνόμια. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε υπόψη τα συμφέροντα των αλλαίων, γιατί τα συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας έχουν αποτύχει παταγωδός στο παρελθόν. Ευχαριστούμε κύριε Χάτον. Το λόγο για τώρα ο κύριος Χάρτον για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε. Ε, είχαμε ακούσει πριν από πολλά χρόνια από το ΠΒΒ ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθουν σε πολύ δυσάρεστη θέση. Βέβαια γελάει καλύτερα όπως γελάει τελευταίος, εμείς δηλαδή. Γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας φαίνεται ότι έδωσε ακόμη περισσότερες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που ήταν μείζον σφάλμα. Στα χωρικά είδατα της Σκοτίας ε, αλλιεύονται αλλιεύεται ρέγγα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καθορίσει τη μέγιστη αλλιευμένη ε, ποσότητα και ε, διαχειρίζεται το απόθεμα. Η προσαρμογή του πολιτού σχεδίου γίνεται πολύ δύσκολη εξαιτία των αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ανήκουστο. Η σημερινή κατάσταση είναι απαράδεκτη. Αν πιστεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα μπορεί να ρυθμίζει τα βιολογικά χαρακτηριστικά μικρών ψαριών όπως η Ρέγγα, νομίζω ότι ε, είναι γελίο. Το κόμμα μου, το PVV, θεωρεί ότι η κοινή ελληνική πολιτική θα πρέπει και πάλι να επιστρέψει στις εθνικές αρμοδιότητες. Για τα κράτη-μέλη είναι σε καλύτερη θέση να διαχειριστούν την αλληλευτική τους πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά. Περνούμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κ. Καντέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Στρούαν Στίβενσον για την έκθεσή του σχετικά με ε, την ε, πολιτική για ε, την Ρέγγα που αυτό θα επηρεάσει τη γενικότερη, το γενικότερο προγραμματισμό για πολλά έτη και ο στόχος τον οποίο θέτουμε θα επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία των επαγγελματιών του χώρου. Την Τρίτη ε, είπαμε ότι ε, πρέπει να... Ε, το Συμβούλιο αρνήθηκε την απαγόρευση των απορρίψεων στη θάλασσα, πράγμα το οποίο είναι πολύ κακό σημάδι διότι προ η πρόταση του Συμβουλίου είναι ε, πολύ επικίνδυνη για το μέλλον της αλληλείας. Εμείς ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία βαθμιαία μείωση των απορρίψεων και ε, η Επιτροπή μας προτείνει να υπάρχουν άδειες που θα μπορούν να μεταφέρονται, αλευτικές άδειες που θα μπορούν να μεταφέρονται ενδιαφέρονται ενώ θεωρώ ότι και εδώ θα πρέπει η διαχείριση της αλληλείας να συνεχίσει όπως είναι τώρα. Δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε τη δραστηριότητα αυτή και σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Μίρσκι στην αίθουσα. Οπότε για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Ντέιβις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 4.30 το πρωί οι Υπουργοί ε, ε, χθες τελείωσαν να συζητούν την ε, αλευτική πολιτική και είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολιετή προγράμματα για κάθε είδο αλίας. Πράγμα το οποίο είναι μια ανοησία εφόσον αντιτίθενται στη δημιουργία αυτών των πολιετών προγραμμάτων το Συμβούλιο θέλει να μπορεί να συνεχίσει, να μπορεί να επιτρέψει στους υπουργούς να θέτουν τις ποσοστώσεις κάθε χρόνο, γιατί είχαν μεγάλη επιτυχία. Κάθε χρόνο το Δεκέμβριο καθόριζαν τις, τους φόρους και τις ε, ποσοστώσεις και γι' αυτό έχουν καταστραφεί ε, τόσο τα αποθέματα τα λιευτικά. Ε, και θέλουν αυτά να περιληφθούν σε μακροπρόθεσμα προγράμματα. Αλλά ξέρουμε τι λένε οι συνθήκες ε, και ξέρουμε ότι υπάρχει μία διαφορά η οποία πρέπει να επιληθεί και μπορεί να επιληθεί η διαφορά με το Συμβούλιο μόνο γύρω από ένα τραπέζι συζητήσεων. Ο κύριος Στίβενσον ζητά την ε, συνδρομή της Κυπριακής Προεδρίας αλλά εγώ προσβλέπω ε, και στις 15 μέρες που έχει ακόμη η Ιδανική Προεδρία να καταρτήσει μία ε, διαδικασία για να μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατόν να εφαρμόσουμε αυτά τα πολιετή προγράμματα για την αλληλευτική πολιτική. Κύριε Ντέιβις, ο κύριος Χάρτονγκ σας ε, απευθύνει μία μπλε κάρτα. Τη δέχεστε. Κύριε Χάρτονγκ, έχετε το λόγο. Αγαπητέ συνάδελφε, ε, διάβασα σε μία Ολλανδική εφημερίδα ότι η Βόρειος Θάλασσα είναι γεμάτη και ξεχυλίζει από ρέγγες και εσείς μας, λέγετε, λέτε ότι μειώνονται τα αλλιευτικά υποθέματα. Αυτό δεν είναι αληθές. Μήπως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το ελέγξει αυτό μέσω ανεξαρτήτων παρατηρητών. Τι γνώμη έχετε. Ευχαριστώ. Σχετικά με την ε, Επιτροπή υπάρχουν 20 ε, ε, αποθέματα τα τα οποία βρίσκονται εις το ανώτατο επίπεδο αποδόσεως ε, πράγμα το οποίο είναι ήδη μία πρόοδος αλλά ε, πιστεύω και μπορεί να με διορθώσει όποιος ξέρει καλύτερα τα πράγματα η Ρέγγα είναι ε, σχετικά σε μία καλύτερη κατάσταση από ότι είναι ο Μπακαλιάρος ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, κύριε Συγητά Στίβενσον. Η σκοτσέζικη ρέγγα έχει μεγάλη επιτυχία ε, στις κάτω χώρες. Ε, βέβαια έχουμε και φρέσκια ρέγγια, αλλά η σκοτσέζικη ρέγγια, τη χάνει μεγάλης επιτυχίας μεταξύ των Ολλανδών καταναλωτών έχει 80% ε, ωφέλιμα λιπαρά και διαπιστώνουμε ότι έχουμε πολύ περισσότερες ρέγγες από ό,τι στο παρελθόν, πολύ περισσότερα θέματα από ό,τι φανταζόμασταν. Έχω λοιπόν ένα μήνυμα. Ε, οι επιστημονικές προβλέψεις θα πρέπει να βελτιωθούν γιατί υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Γι' αυτό καλό θα ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιμείνει να έχει λόγο και να μην αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει μόνη της αποφάσεις. Πρόκειται για εξουσίες και αρμοδιότητες που κατοχυρώνονται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ίδια τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα πρέπει να τις διεκδικήσουμε αυτές τις εξουσίες, να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πολύ σωστή ήταν η προσέγγιση του εισηγητού μας του κυρίου Στίβενσον. Θα πρέπει απλώς να μπορούμε να επιμείνουμε προασπίζοντας τα, δικαιώματά μας είναι επιτέλους ε, καιρός να ε, ακούσουμε και να ακουστεί και η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye. Δύο ζήτησαν το λόγο στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής. Ο πρώτος είναι ο κύριος Σον Κέλλη. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω τέτοιες ε, εμβριθείς γνώσεις για τα αλληλευτικά αποθέματα όπως η κυρία Πάτε Κόπ Κάλαχαρ και Στρούαν Στίβενσον αλλά και στην δική μου πατρίδα έχουμε ανεπτυγμένη αλληλεία γι' αυτό και με ενδιαφέρει η συζήτηση αυτή μερικά από τα σχόλια που άκουσα πραγματικά με... μου δημιούργησαν φοβερή δυσφορία και δυσανασχέτηση. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για την Αλία, αλλά είναι κάπως απογοητευτικό ε, να, λέμε, να ακούμε ότι η έκθεση έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο, όχι μόνο η έκθεση του κυρίου Στίβενσον, αλλά και η έκθεση του κυρίου Γκάλεχερ. Είναι απαράδεκτο αυτό το διέξοδο και το μπλοκάρισμα που έχει δημιουργηθεί στο Συμβούλιο. Και το πνεύμα και το γράμμα τη συνθήκη τη Λισαβόνα θα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Και σίγουρα εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μα και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μα. Έχουμε ένα τεράστιο χρέο για την απέναντι στην Αλία και στου Αλεί. Θα πρέπει λοιπόν να ευοδοθούν αυτά τα πολιτή σχέδια διαχείριση ελεία. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, όπω είναι και οι απορρίψει. Και προσβλέπουμε στι δύο διαδοχικέ προεδρίε, την Κυπριακή και την Ιρλανδική, να φέρουν σε αίσιο πέρασα αυτή τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Γκαμπριέλ Αντρόβερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλούμε για ρέγγες, μιλούμε για πολυετή σχέδια διαχείρισης αποθεμάτων, αλλά κυρίως μιλούμε για δικαιοδοσίες, για αρμοδιότητες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαιώματα αρμοδιότητες. Θα πρέπει ε, και το Συμβούλιο να σεβαστεί και να εφαρμόσει τη συνθήκη της Λισαβόνας και επιπλέον να σεβαστεί και τη γνώμη των νομικών υπηρεσιών έχουμε συναπόφαση και μια πολιτική απόφαση του Συμβουλίου όχι μόνο κατά στρατηγή της αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που δεν πρέπει ούτε θα δυνάμεθα να δεχτούμε, αλλά διακυβεύει και πολύ σημαντικά ζητήματα με τη στάση του Συμβουλίου όπως είναι η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Απευθύνομαι στον απόντα εκπρόσωπο του Συμβουλίου και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήματα είναι πολύ πιο σοβαρά από, από όσο αντιμετωπίζονται από το Συμβούλιο. Παρακαλώ να το λάβετε υπόψη. Ευχαριστώ. Το λόγο και τώρα ο Επίτροπος Ντάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη για τη συμβολή τους στη συζήτηση αυτή. Αυτό δείχνει ότι το Κοινοβούλιο ε, παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να ε, καθησυχάσω τους βουλευτές ε, ότι πραγματικά η Κομισιόν εξεκολουθεί να προσπαθεί ε, να λύσει το θέμα των πολιετών ε, προγραμματισμών με το Συμβούλιο. Το σημαντικό είναι να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, ότι πρέπει μάλλον να προχωρήσουμε με αυτά τα εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την βιώσιμη αλληλεία. Ευχαριστώ πολύ. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση θα δώσω τον ε, λόγο ξανά στον εισηγητή κύριο Στίβενσον. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο κύριο Στίβενσον. Λυσμονήσατε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Ντάλη αλλά και όλους τους ε, συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Επανειλημμένα ακούσαμε από τους ε, συναδέλφους που πήραν το λόγο ε, ότι το κύριο πρόβλημα, το κύριο ζήτημα είναι το μπλοκάρισμα των πολιετών προγραμματισμών από το Συμβούλιο. Τα θέματα είναι τόσο σημαντικά που η Επιτροπή μας υπό τον Γκαμπριέλ Μάτο ε, πήγε να συναντήσει την Επιτροπή και είπε για μία ακόμα φορά ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει σαν ε, κύρια προτεραιότητα τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε οι άμεσα εκλεγμένοι, εμείς είμαστε ε, οι δημοκρατικά εκλεγμένοι. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν και δυστυχώς δεν έχουμε ούτε καν εκπρόσωπο της δανικής προεδρίας δεν, δεν είχαν ε, καν την, δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να ούτε καν να ακούσουν, να παρακολουθήσουν τη συζήτηση αυτή. Βεβαίω θα συζητηθεί το θέμα με την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία αλλά ε, θα το συζητήσουμε και με τον ίδιο τον πρόεδρο Βαν Ρόμποϊ ε, γιατί πραγματικά πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να δείξω και ένα τελευταίο ζήτημα. Κύριε Επίτροπε Νταλή, είπατε ότι δέχεστε και σας είμαι ευγνώμων τις περισσότερες τροπολογίες της έκθεσής μου. Αλλά σας ε, προβληματίζει λίγο ότι όταν ζητούμε ε, την ε, όταν λέτε ότι θα πρέπει να διαβουλευτούμε με την με τους εμπλεκόμενους φορείς It's avoiding consultation with the stakeholders that has led και με το ΕΑ και με το Συμβούλιο των to look carefully at the result of today's vote το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των Πελεγωγικών Ειδών. Σας προβληματίζει αυτό, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ολοκληρωθεί η συζήτηση λοιπόν και για το θέμα αυτό. Ψηφοφορία δεν θα λάβει χώρα στις 12 σήμερα. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μερισίας διατάξεως. Η αφορά δήλωση της Επιτροπής ε, σχετικά με τους Ευρωπαίους παραγωγούς γάλακτος.